Την ε, Τετάρτη θα υπογράψω 16 τέτοιες ε, πράξεις σύμφωνα με τον κανόνα 74 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Οι τίτλοι των πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Και υπάρχουν επίσης ε, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα περνάω στις αλλαγές της ημερησίας διάταξης η τελική ημερήσια